Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Καλώς ήρθατε συνάδελφοι, καλώς ήρθατε καλεσμένοι από το Συμβούλιο, την Επιτροπή. Καλώς ήρθατε βοηθοί, εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων και φορέων που λαμβάνουν μέρος σήμερα και παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε διερμηνείς υπάρχουν παρατηρήσεις για την σε διάταξη. Η κυρία Χάζεκαμπ. Eh, eh, Ευχαριστώ. Πριν ψηφίσουμε, να αναφερθώ σε κάτι διαδικαστικό. Χρειάζεται πολιτική απόφαση να μην ψηφίσουμε τις τροπολογίες όταν κάποια άρθρα βρίσκονται συμβαστικές. Οι τροπολογίες μάλλον που δεν είναι εντός των συμβαστικών. Ζητώ σε κάθε περίπτωση στις τροπολογίες 38, 39 και μια άλλη να ψηφίσουμε. Οι συμβαστικές τροπολογίες καλύπτουν ε, αρκετές τροπολογίες, αλλά καλό θα ήταν, μια και το θέσατε, να το ελέγχουμε κάθε φορά ποιες τροπολογίες καλύπτει κάθε συμβαστική πρόταση. Κανονικά τις καλύπτει όλες, αλλά αφού το ζητήσετε θα το ελέγχουμε κάθε φορά ότι στιγμή δηλαδή που θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη συμβαστική τροπολογία. Η ε, κυρία Ζωανά. Τεχνικό πρόβλημα έχω, ξέρετε. Η διερμηνία, κάτι με το κανάλι δεν δουλεύει. Δεν ακούω τη διερμηνία. Τεχνικό είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν καταλαβαίνω τα πολωνικά. Μήπως αναλάζετε θέση. Όχι, τίποτα δεν ακούω. Ε, αλλάξτε θέση τότε. Nie mamy nikogo. No, no, δεν βλέπω κανένα στην ρουμανική καμπίνα. Μήπω δεν έχει διερμηνία. Θα πρέπει να βολευτείτε με τα αγγλικά. Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανείς στη ρουμανική καμπίνα σαν να βάλουμε την ψηφοφορία. Yes, I know. Το ξέρω. Κυρία Ζανά, παρακαλώ, ακούστε αγγλικά. Ακούστε την αγγλική καμπίνα. Ε, εντάξει, με τα γαλλικά θα πορευτώ. Αρκεί για μένα. Μάλιστα, ανακοινώσει. Ο κύριος Χόισλινγκ κάλεσε δημοσιογράφους από το κρατικό κανάλι Τσεντεφ παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες. Δεν έχουμε δηλαδή και ρουμανικά μεταξύ άλλων. Κανονικά ρουμανικά έπρεπε να είχαμε, δεν ξέρω τι συνέβη. Πάμε στο σημείο 3 τώρα. Που είναι το κυρίως θέμα. Τα στρατηγικά σχέδια τη κοινή γεωρικής πολιτική, στα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών. Η συγγήτρια, όπως όλοι γνωρίζουμε για την έκθεση αυτή, είναι η κυρία Έστερ Ράν Γκαρσία. Και πολλέ επιτροπέ η ΔΕΒΕ, ΙΝΤΑ, προπολογισμών, ελέγχου προπολογισμού ΕΜΒΙΤΡΕ, ΡΕΤΖΙ και γυναικών έχουν συντάξει γνωμοδοτήσεις επί της εκθέσεως της κυρίας Γκαρσία. Σήμερα θα ψηφίσουμε τρεις ε, μία από τις τρεις ε, εκθέσεις του πακέτου. Χθε ψηφίσαμε μία. Έχουμε 5.253 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, 448 από την εισηγήτρια, 670 τροπολογίες από τις επιτροπές που έχουν νομοδοτήσει, 201 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, που είναι συνδεδεμένη επιτροπή δυνάμει το άρθρο 54 με κοινέ αρμοδιότητες. 124 συμβαστικές τροπολογίες καλύπτουν 110 άρθρα και 3 παραρτήματα, εκ των οποίων 10 Εναλλακτικέ τροπολογίε έχουν κατατεθεί για το άρθρο 9 και μία για το παράρτημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλου που ε, συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτή τη έκθεση και την επεξεργασία των τροπολογιών, την εισηγήτρια, τους σκιώδης τους βοηθούς τους, συνεργάτε τους, τη γραμματεία και σίγουρα θα προτείνουμε και κάποια διαλύματα. Το, πρώτο θα γίνει πριν την ψηφοφορία της συμβαστικής, έκθεσης, της συμβαστικής τροπολογίας για το άρθρο 91 και μετά την τελευταία τροπολογία για το άρθρο 90 και θα διακόψουμε στις 12.30 και θα ξαναρχίσουμε στις 2.30 για τη συνέχιση των τροπολογιών και της ψηφοφορίας. Επειδή δεν έχουν εξεταστεί όλες οι τροπολογίες από τους γλωσσομαθείς νομικούς, θα πρέπει μετά το τέλος της ψηφοφορίας να γίνει διόρθωση ή ε, από τη σκοπιά των ε, γλωσσομαθών νομικών προκειμένου να γίνει συμβατή διατύπωση και να αποφύγουμε τις αντιφάσεις. Το ίδιο και για, την για τις αιτιολογικές σκέψεις θα γίνει εξέταση του κειμένου προκειμένου να αποφευθούν οι αντιφάσεις, να εξασφαλιστεί μια συνοχή του κειμένου. Και αυτό θα γίνει με τη συνεργασία της Γραμματείας ε, και των γλωσσομαθονομικών, ώστε το αιτιολογικό να συμβαδίζει με το διατακτικό. Θα ψηφίσουμε με τους συνήθεις κανόνες, κανονικά διανατάσσεως της χειρός. Έχουμε όμως και πολλές συμβαστικές τροπολογίες, ε, ονομαστικές τροπολογίες και κάθε συμβαστική τροπολογία καλύπτει το σύνολο του συγκεκριμένου άρθρου. Οπότε σε περίπτωση που γίνει δεκτή συμβαστική τροπολογία, καταπίπτουν όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες που αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο. Ακόμη και αυτές που προτείνουν προσθήκες ε, υποσημείων ή συμπληρωματικών παραγράφων μόνο οι τροπολογίες που δεν καλύπτουν από συμβαστική τροπολογία και που δεν είναι αντιφατικές με αυτή θα τεθούν στη συνέχεια σε ψηφοφορία. Η συγγετρία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τις άοκνες προσπάθειες τους και τη συνεργασία. Να ευχαριστήσω θερμά τους και οδησηγητές των πολιτικών ομάδων γιατί ήταν πολύ σημαντική η συνεργασία μας. Και να ευχαριστήσω και τους συντάκτες γνωμοδότης και τους σκιώδεις συγητές των γνωμοδοτήσεων, γιατί έχουμε ένα πακέτο νομοθετικών μεταρρυθμίσεων. Η έκθεση μου είναι μία από τις εκθέσεις αυτού του πακέτου. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και στα υπόλοιπα πακέτα. Χθε ψηφίσαμε για την ενία κοινή οργάνωση αγορών, την έκθεση του κ. Ατρίου. Σήμερα ψηφίζουμε τη δική μου έκθεση, που ίσω είναι και οι πιο δύσκολη τα στρατηγικά σχέδια. Και ευχαριστώ θερμότατα και τη γραμματεία που ήταν ε, εξαιρετική στην συνεργασία και ανεκτήμητη συνεισφορά της. Όπως είπε και χθε ο κύριος Αντριέ, το έργο αυτό έγινε με αρκετή πίεση χρόνου, γιατί είμαστε στο τέλος της θητείας και μας ε, υπευλήθη σχετικά καθυστερημένα το έγγραφο μετά την ε, καθυστερημένη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη δική μου πολιτική ομάδα, γιατί χωρίς την στενή συνεργασία και την ε, αμέριστη υποστήριξη της πολιτικής μου ομάδας δεν θα ήμουν σε θέση να διεκπαιρεώσω το έργο μου. Επίσης να ευχαριστήσω τις γραμματείς και των πολιτικών ομάδων και κυρίως της δικής μου πολιτικής ομάδας για την ανεκτήμητη προσφορά τους. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τους τέσσερις συνεργάτες μου, τη Γιολάντα, τον Αρτούρο, τον Νταβίτ και τη Μαριανέλα. η βοηθοί μου αφιέρωσαν όλες τις ελεύθερες του στιγμές, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, τις αργίες, τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους. Τησίασαν τα πάντα και μας επέτρεψαν να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για να δούμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής Γεωργίας για το θέμα αυτό, γιατί ζητούμενο είναι το συμφέρον των γεωργών και των τρόφων και πάνω απ' όλα το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η ΚΑΠ έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ποιοτικά τρόφιμα σε προσιτές τιμές για όλους τους Ευρωπαίους. Οπότε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία. Θα ευχαριστήσουμε και στη συνέχεια τους συντελεστές αυτής της έκθεσης. Πάντως, όπως είπατε, όλοι οι γεωργικοί κτηνοτρόφοι, αλλά και οι συμπολίτες μας έχουν στραμμένα τα μάτια τους σε εμά και περιμένουν την έκβαση του έργου μας. Ο κύριος Αλμπερντέσιτσε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λόγω τη αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού πρόσφατα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποσύρω το όνομά μου από, από την τροπολογία 449. Αποσύρω τη συγκεκριμένη τροπολογία και το όνομά μου. Σα ευχαριστώ. Αποσύρετε σχετική τροπολογία. Ο κύριο Ταραμπέλα ζήτησε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομο διότι το εξήγησε στην προηγούμενη συνεδρίαση γιατί ε, έχω προτείνει αυτή την ε, τροπολογία, αυτή την απόρριψη. Μόνο περιθωριακά μπορεί να βελτιωθεί ε, το κείμενο. Δεν μπορούμε να αναδιτυπώνουμε το κείμενο κάθε πέντε χρόνια. Αναμφισβήτητα έκανε δουλειά ο εισηγητής και όλοι οι εισηγητές. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί σεβασμό. Γι' αυτό θα μείνω για να για να ψηφίσω, διότι ελπίζω ότι η απόρριψη δεν θα έχει πλειοψηφία. Στο τέλος, θα δούμε ότι με την τροπολογία δεν θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση. Εγώ επιμένω στην απόρριψη και ε, υποστηρίζω εν ονόματί μου και την τροπολογία του κυρίου Ντέσ, όπως είπα πριν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ταραμπέλα ανέλαβε την τροπολογία του κύριου Ντές και επιμένει στην κατάθεση της. Υπάρχουν ερωτήσεις μήπως, απορίες? Όχι. Έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, οπότε θα ψηφίσουμε Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία του κυρίου Ταραμπέλα, δηλαδή υπέρ της απόρριψης της θέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. E Έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Okay. W Ψηφίσατε όλοι. Μπορώ να κλείσω την ψηφοφορία. Ωραία, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία ταραμπέλα. Με 10 ψήφους υπέρ και 29 κατά. Οπότε, μια και δεν αποδόθηκε η απόρριψη της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ψηφίζουμε κανονικά την έκθεση. Διανατάσσω στις χειρός καταρχήν και αν χρειαστεί τίποτα άλλο θα το πούμε. 451 τροπολογία του κυρίου Χόισλινγκ. Χόιμπουχ και άλλοι. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Πρώτη της Δεύη υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 450 υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 2. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 1091. 1091. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1093 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1094 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1094. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 1095 υπέρ. 1095. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1096 υπέρ. Εγκρίνεται. Ε, θα ψηφίσουμε μαζί τρεις τροπολογίες. Τη 1097, τη 1101 και 54 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 1098 και 53 της ΕΜΒ υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 1099 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1100. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1100. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1102 και 55. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 1103. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Εγκρίνεται. 1104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 1104. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 1105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 49 και 1107. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 1108 του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1109 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 4. Πάλι με ονομαστική κλίση. Άρχεται η, συμβαστική, η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 4. Ονομαστικά. Τέλος. εγκρίνεται. Πάμε στη συμβεστική 5-6. Είναι αρκετές σελίδες παρακάτω και χαιρόμαστε γι' αυτό ότι κερδίζουμε. Σε μένα είναι στη 13 σελίδα, δεν ξέρω στη δική σελίδα, 5-6 συμβαστική τροπολογία με ονομαστική κλίση, άρκετη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Ο κύριος Άγνιος ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που αναφέρατε την αριθμό της σελίδας. Βοηθάει. Αν συνεχίσετε να λέτε τον αριθμό της σελίδας, καταλαβαίνω ότι όσο περνάει η ώρα, ίσως κάπως να μας ξεφεύγουν οι σελίδες, ανάλογα, να αλλάζει η σειρά των σελίδων, ανάλογα με την κατάσταση ψηφοφορίας, αλλά μας δίνει μια ιδέα τον, τον αριθμό. Γυρίζουμε μια σελίδα, 7 σελίδες. Ευχαριστώ. Θα λέω τον αριθμό των σελίδων, τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ μπροστά μου και υπολογίστε εσείς. 1508 στη σελίδα 24. Σελίδα 24. Στη σελίδα 24 πάμε και στην τροπολογία 1508. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1508 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση ή όχι. Α, συγγνώμη, ξέχασα την 51 της ΔΕΒΕ. Ψηφίζουμε την 51 της ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Οπότε τώρα περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην επόμενη συμβαστική τροπολογία. Πάλι με ονομαστική κλίση. Συμβαστική τροπολογία 8. Μία σελίδα παρακάτω. Άρχιτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 9, ονομαστική ψηφοφορία και εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 1567. Στη σελίδα 27. 1567 του κυρίου Χόισλιν και άλλων. Θα Αναφέρω και το όνομα του συντάκτη τη τροπολογία, γιατί είναι πιο εύκολο να βρείτε έτσι την τροπολογία. 1567 Χόισλινγκ. Ποιο είναι υπέρ. Μαζί με την 69 τη Ρέτζη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 64 τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Υπέρ. Εγκρίνεται. 65 τη ΕΜΒ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1568 και 70. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 53 της ΔΕΒΕ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1569 και 66, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 10, 10. Πάλι υπεράριθμοι στο ΕΛΚ. Ψηφίζουν περισσότεροι από ό,τι δικαιούνται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία, η συμβαστική 10. Πάμε στην 1586 τώρα, τροπολογία 1586, στην ίδια σελίδα, την 28. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας Hoisling και λοιπόν, υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογίες 52 της ΔΕΒΕ και 67 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία... Συμβαστική τροπολογία 11 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ονομαστικά. Στη σελίδα 30. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 12. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη σελίδα 34 και στην τροπολογία 1700. 1700 τροπολογία, σελίδα 34. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13, με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 1797 τώρα, στη σελίδα 39 του καταλόγου ψηφοφορίας. Τροπολογία 1797 στη σελίδα 39 της κυρίας Χόιμπουχ και του κυρίου Ροπέ είναι η σχετική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1796. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1795. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1824 της κυρίας Άνερα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1798 της κυρίας Ένρα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70 τροπολογία 1799 του κυρίου Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1800 Νόιχλ και Ταραμπέλα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 1800. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1802 του κ. Χόισλιν και άλλων. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1803 Νόιχλ και άλλων. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1801. Τα 1805, συγγνώμη, λένε και άλλο. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1800 νόηχλου και λοιπόν, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1806, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 1807. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1808 και 1809. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 1810. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1811. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1812 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1813 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1814 υπέρ. Εγκρίνεται. 1815 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο για τροπολογία 1815 άρχεται η ψηφοφορία. 1815 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 1816. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 1817. Υπέρ εγκρίνεται. 1818 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1819 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1820 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1822 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1823 υπέρ, εγκρίνεται. 57. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1823. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπερδεύτηκε η κυρία Νάχλη γιατί ψήφισε υπέρ με το χεράκι της. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 57 της ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 73 της ΕΜΒΗ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. οπότε περνάμε στην τροπολογία 2006 στη σελίδα 50 πάμε στη σελίδα 50 Ω, σας ευχαριστώ γιατί Περάσαμε πολλές σελίδες. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2006. Κυρία Μαγκίνε ζήτησε το λόγο. Στο συγγνώμη που διακόπτω. Για αυτή την τροπολογία η λέξη έχει διαγραφεί ο ενεργός, ο ε, καλλιεργητής, έχει, ο αγρότης έχει διαγραφεί και αναγράφεται μόνο αναγράφεται η λέξη αγρότης αντί ενεργό αγρότης. Υπάρχει διαφορά στον ορισμό. Ίσως μπορούμε νομικά να το εξετάσουμε μετά την ψηφοφορία και να το ξεχνιάσουμε αυτό. Καλό σίγουρα θα ελεγχθεί από τους γλωσσομαθείς νομικού. Σας ευχαριστούμε για την παρατήρηση κύριε Μακίνε. Και ψηφίζουμε τη 2006 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2006. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 102 και 103. Ποιος είναι υπέρ, μαζί τις ψηφίζουμε, τη ηγήτριας είναι υπέρ, εγκρίνονται. Τροπολογίες 104 ή μάλλον πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 102 και 103 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται τελικά. Εγκρίνονται, λέει ο πρόεδρο. Όχι, όχι, λάθο, λάθο. Απορρίπτονται, απορρίπτονται. Από την αριστερά ποιο είναι ο συντονιστή. Γιατί. Α, η κυρία Νόχλα, εντάξει, θα με βοηθήσει στην καταμέτρηση. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Με βοηθάει να ξέρω ποιο συντονίζει. Τροπολογίες 104 και 2009 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 105. Προηγουμένως όμως θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά τις τροπολογίες 104 και 2009 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνονται. Τροπολογία 105 της συγγήτριας. και της κυρίας Αγγιλέρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 105 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Odrzucona. Απορρίπτονται. Τροπολογία 2011. Α, ε, συγγνώμη, 2010. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 2012. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2012 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 106. Έχουμε προφορική τροπολογία εδώ. Ποιος θα την υποβάλει. Η κυρία Ερνάς Γκαρσία. Τη βλέπετε στα σχόλια την προφορική τροπολογία, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Καλώς. Ποιος είναι υπέρ της 106. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2013 ή μάλλον 2014 2014 του κυρίου Νταντάν, λέει ο πρόεδρος. Όχι, 2013 πάλι, λάθος κάναμε. 2013. We are going to 83. Όχι, λάθος λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην 83 της Ρέγγι. 83 Ρέγγι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2021. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2021. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Ο Τζουτσόνα. Απορρίπτεται. 107 της ηγήτριας. Ή μάλλον 2022 πρώτα, διορθώνει ο πρόεδρος, του κυρίου Μπιτσότο. 2022, ποιος είναι υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 107 της ηγητρίας, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2025 του κυρίου Φλάναγκαν. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ε, μάλλον, μάλλον πάμε στην 2023 ε, κατευθείαν. 2023, Όζου, Κούσμιου, Κοσιεύσκα κτλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία για τη 2023 και λοιπές μαζί. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 2029. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 108. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 2030. Ποιος είναι υπέρ. ή μάλλον λάθος, λάθος. 2033, στη μεθεπόμενη. Τη κυρίας Αγγιλέρα είναι και αυτή, αλλά η επόμενη. Ποιο είναι υπέρ, 233. 2033. Εγκρίνεται. Πάμε στην 109 της συγγήτριας. 109 και 2031 και 32. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα την 2034. Ε, Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 2036. Νοίχλ, Ταραμπέλα και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2037. Νόιχλ και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2037 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 2038 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2039 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2040 υπέρ. Εγκρίνεται. 2041 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2042 και άλλες. 43, 44 κλπ. Υπέρ. Εγκρίνονται. 2047 ή μάλλον όχι, πρώτα τη 2046 του ε, κ. Ερντός υπέρ, Όχι, λάθος. Επανερχόμαστε στη 2047. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2049 και 76 εμβι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 2048 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 19. Με ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20, στην επόμενη σελίδα. Ή όχι. Όχι. Πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε την εναλλακτική. Εναλλακτική συμβαστική τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία Ρας Γκαρσία. Εμένα άλλα λέει ο κατάλογος ψηφοφορίας. Μου λέει ότι μετά την συμβαστική τροπολογία 19 θα πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα τη συμβαστική τροπολογία 20. Ή κάνω λάθος. Όχι. Πρώτα την εναλλακτική συμβαστική πρέπει να ψηφίσουμε, μου λέει η γραμματεία. Ο κύριο Άγνιο. Πρόεδρε, ίσως δεν κατάλαβα καλά. Αλλά η συμβαστική ψηφοφορία ήταν αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο ψηφοφορίες για συμβιβαστική. Για ποια συμβιβαστική μιλάμε. Θα ψηφίσουμε την εναλλακτική συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 με ονομαστική κλίση. Είναι ακριβώς στην επόμενη σελίδα. Εναλλακτική συμβαστική τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 2911, στη σελίδα 56 του κυρίου Ντόρφμαν, 2111. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2114. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2114, 2114. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2115. 2115. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2116 του κύριου Κάρθη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως καλύτερα για την 2116, μια και το ζητήσατε. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστικές τροπολογίες 22 και 23 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνονται. Τροπολογία 2144 στη σελίδα 58 του καταλόγου. Πρόκειται για τροπολογία Ντόρφμαν και Κάρθη που είναι πανομοιότυπη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 2146, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 2149, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 29.47 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 21.48 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 21.50 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2150 του κ. Γιάρα, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το ξέρω, το ξέρω. 21.59 το, 51, ε, το κύριο Νταντά υπέρ. Εγκρίνεται. 21-52, Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τροπολογία 21.52. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 25, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 26, στην σελίδα 60. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 26. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 27 στη σελίδα 63 του καταλόγου ψηφοφορίας. Συμβαστική 27. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη σελίδα 65 και στην τροπολογία 2276 της κυρίας Αγγιλέρα. 2276. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 83 έμβη, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2277. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 2278 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2279 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 28 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 2472, στη σελίδα 74, τροπολογία 2472 στη σελίδα 74. Χαίτεμα και άλλων. 2472. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2931, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Και πάμε στην τροπολογία 2556 στη σελίδα 78. Τροπολογία 2556 της κυρίας Χόιμπουχ. Μαζί με την 94 έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 2557 και 2558. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογίες 25-59 και άλλες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τροπολογία 2563. 63. Ποιος είναι υπέρ. Πού πάτε. «2570». Πάμε στην 2570 της κυρίας Γκοσεύσκα. 2570 και 2571 υπέρ εγκρίνονται ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες Γκοσεύκα, Γκοσεύσκα και Γιάρντες και τα λοιπά. Μαζί 2570 και 2571. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνονται. Τροπολογία 2572 και 95 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 2573 του κυρίου Νέκοφ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2574 του Νέκοφ και πάλι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 150 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 151 της ηγετρίας υπέρ. Εγκρίνεται. 151, 152 ε, της ηγετρίας υπέρ. Εγκρίνεται. 153 της ηγετρίας υπέρ. Εγκρίνεται. 2575 της κυρίας Αγγιλέρα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 2575. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 2576 του κυρίου Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάει ο ένας κατάλογος. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα ή δεν χρειάζεται. Αργότερα. Καλώς. Οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 39 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Ονομαστικά για την συμβαστική 40. Τέλος ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 41. Συμβαστική 41 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 42 στην επόμενη σελίδα, σελίδα 3, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 43, σελίς 5. Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. 43 συμβαστική τροπολογία. 43 με ονομαστική κλίση, συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 44 στη σελίδα 10. Με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ένας υπεράριθμος από το ECR. εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 2806 στη σελίδα 12 του καταλόγου ψηφοφορίας. Τροπολογία Αγγιλέρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2807 Σράιερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2808 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2809 υπέρ. Εγκρίνεται. 28-12 της κυρίας Σράιερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28-13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28-14 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28-15 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 2815. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 46 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία για τη συμβαστική 46. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 2866, Λίνς, στη σελίδα 15. 2866, Λίνς, Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2864, Ερντός. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 2864, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2865. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 2867 και 2868. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 2869 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2870 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστικές τροπολογίες 48 έως 50 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για τις συμβαστικές 48-49-50. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 51 σελίδα 19. Συμβαστική 51 στη σελίδα 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Με ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 52. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Είναι στη σελίδα 21 η συμβαστική αυτή τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Συμβαστική 52. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 53 στη σελίδα 24 στο δικό μου κατάλογο με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 54 στη σελίδα 25 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 54 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 118 της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη σελίδα 26. Έμβη 118 Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογίες 3070 και 3071 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 30, 72, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3072, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 119α της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3073 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3074 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Sprawdzamy, sprawdzamy, głosujemy. Zamykam głosowanie. Απορρίπτεται. 3075 Νταντάμ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 119 Β τη ΕΜΒΗ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3076. Ποιο είναι υπέρ εγκρίνεται. 230 η ηγήτρες υπέρ, εγκρίνεται. 3077 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 231 της συγγήτριας, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 3078 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 3079 και 119 δέλτα υπέρ, εγκρίνονται. 3086. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3086 άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3087. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 120 εμβοί. υπερ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. υπερ υπέρ. Εγκρίνεται. υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30-82 και 83-84 υπέρ. Εγκρίνονται. 30-85 υπέρ. Εγκρίνεται. 30-88 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 30-89 υπέρ. Εγκρίνεται. 30-90. Ή μάλλον 30-91 της κυρίας Εράς 3091 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3091. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30-92, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30-94, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. υπέρ. Α, μάλλον 30-96, λάθος. 30-96, του κ. Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 30-97 υπέρ. Εγκρίνεται. 30-98 και 121 της έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 63 της ΔΕΒΕ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 122 έμβη και 30-99 Χόισλεν και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Συμβαστικές τροπολογίες 59, 60, 61, 62 και 63 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Και πάμε στη τροπολογία 3255, στη σελίδα 37. Τροπολογία 3255. του κυρίου Ντες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 64 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 65, στη σελίδα 39, με ονομαστική κλίση. Συμβαστική τροπολογία 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 66, στη σελίδα 46. Σελίδα 46. Συμβαστική τροπολογία 66. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 67. Στη σελίδα 47. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Ονομαστική ψηφοφορία για τη συμβαστική 67. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 68, σελίδα 48. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την συμβαστική 68. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 68α. 68α συμβαστική με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 69. Ή ε, μάλλον 68. Όχι λάθος, λέει ο πρόεδρος. Σελίδα 55, 68η, σελίδα 55, 28β, συγγνώμη, με ονομαστική κλίση, συμβαστική 68β, σελίδα 55, τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 69, συμβαστική τροπολογία 69, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική 69. Και πάμε στην τροπολογία 3666 στη σελίδα 59. Ή μάλλον, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, αργότερα. 69 με ονομαστική κλίση, συμβαστική 69 με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία 70, στη σελίδα 59, σελίδα 59, συμβαστική τροπολογία 70, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 3763 3763 στη σελίδα 63. Ψηφίζουμε την 3763. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 71 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 37, 95. 37 σελίδα 65, πρόκειται για τροπολογία της κυρίας Εράνς και άλλων. 37-95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 38-24 και 38-25. Ποιος είναι υπέρ ή μάλλον λάθος, λάθος. Πάμε στην τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 72 με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 3822 τροπολογία, στην επόμενη σελίδα. 3822 του κυρίου Τόρες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Τροπολογία 38, 23 και 124 της Ρέτζη. Υπέρ. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 72α. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 72α συμβαστική τροπολογία. Εγκρίνεται. Και πάμε στις συμβαστικές τροπολογίες 73 έως 78 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία για τις συμβαστικές τροπολογίες 73 έως 78. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Κυρία Χάζενκαμπ. Εγκρίνονται κυρία Χάζενκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Αν η γραμματεία ε, μπορεί να το ελέγξει παρακαλώ. Τι ψηφίσαμε τελικά. Μέχρι την 78. Μήπως να ψηφίσουμε ξεχωριστά 3, 8, 7, 8. Παρακαλώ. Σταυρομαχίες. Mm. Την 3878 είπατε Η γραμματεία μου λέει ότι δεν γίνεται να ψηφίσουμε για την 3878. Λυπούμε κυρία Χάζεκαμπ. Αλλά αυτά προβλέπει η διαδικασία. Οπότε περνάμε σε ποια συμβαστική την 79. Όχι, προηγείται η συμβαστική τροπολογία, εναλλακτική συμβαστική τροπολογία 7. Εναλλακτική συμβαστική 7, στη σελίδα 70. Συμβαστική τροπολογία, εναλλακτική συμβαστική 7, στη σελίδα 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 79 τώρα. 79 συμβαστική τροπολογία. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Συμβαστική 79. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 80. Με ονομαστική κλίση και αυτή. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 81 στη σελίδα 71. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 82, λίγο πιο κάτω. Με ονομαστική κλίση Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 83, σελίδα 72. Συμβαστική τροπολογία 83, με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 3915 στην επόμενη σελίδα. Πρόκειται για τροπολογία του κυρίου Χόισλινγκ, 3915. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 3915, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 85 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 86, στη σελίδα 76. Συμβαστική 86, άρχεται ψηφοφορία, με ονομαστική κλίση. Σελίδα 76, συμβαστική 86, Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία 41-42 στη σελίδα 84 41-42 τροπολογία στη σελίδα 84 Πρόκειται για τροπολογία του κυρίου Ντες, 41-42. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα, εναλλακτική συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 9. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εναλλακτική συμβαστική 9. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 87. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία της συμβαστικής 87. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 4179, στη σελίδα 86. Τροπολογία 4179, Χαίτεμα και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 4179. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 88 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 89. Λίγο πιο κάτω. Με ονομαστική κλίση. Συμβαστική 89. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 90. Συμβαστική τροπολογία 90 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η γραμματεία μου λέει να κάνουμε διάλειμμα. Εσείς τι γνώμη έχετε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Συμφωνούμε όλοι. Πολύ ωραία. Ο κύριος Καλινόφσκι λέει καλύτερα όχι, αλλά η πλειοψηφία λέει ναι. Τελείωσε το διάλειμμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με το τρίτο τμήμα. Καθίσατε όλοι. Ο κύριος Ντες που είναι. Ο κύριος Μπούντα επίσης που είναι. Ψηφίζουμε την συμβαστική 91 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 91 με ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 92. Στην επόμενη σελίδα. Ας περιμένουμε να ψηφίσουν όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία τώρα για τη συμβαστική τροπολογία 92 με ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 42.51 στην επόμενη σελίδα, τη σελίδα 3. Τροπολογία 42.51. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 93. Με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 94 και πάλι ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 94. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 95 τώρα, σελίδα 7. Στην σελίδα 7, συμβαστική τροπολογία 95 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 96 στη σελίδα 8 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 97 στην σελίδα 10 με ονομαστική κλίση Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 97. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 98. Σελίδα 11. Στην επόμενη σελίδα δηλαδή. Με ονομαστική κλίση και αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 98 με ονομαστική κλίση. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 99, σελίδα 12. Με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 100. Η 99 έγινε δεκτή. Στη σελίδα 13. Με ονομαστική κλίση. Συμβαστική τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 44-13, σελίδα 14. Αυτό δεν είπα κι εγώ. 44-13. Τροπολογία Αγγιλέρα. Στη σελίδα 14. Προφορική τροπολογία της κυρίας Αγγιλέρα. Παρακαλώ. Η προφορική τροπολογία συνίσταται στην προσθήκη στον τίτλο για τα προγράμματα περιφερειακής παρέμβασης. Προσθέτουμε λοιπόν στον τίτλο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό προσθέτουμε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου for the Rural Development. Προσθέτουμε στον τίτλο. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Για τη 4413. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4559. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 167 της Ρέτζη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 102 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 103 στη σελίδα 15. 103 με ονομαστική κλίση, συμβαστική τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 104, στη σελίδα 16, επίσημη ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 104. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 4453, 4453, 4454 και 4455 ή μάλλον όχι, λέει ο πρόεδρο λάθος. Μόνο τη 4453 και 4454 ψηφίζουμε μαζί. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για τις τροπολογίες 4453 και 54 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία Εγκρίνονται. τραπολογια 4455, 44-55 έρντας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 4455 55 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. δεν πρόλαβε να ψηφίσει ο κύριος Δεκάστρο. Μπράβο κυρία Αγγιλέρα. Ε, μήπως θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ε, ναι, αλλά πήρατε καφέ. 106. Συμβαστική τροπολογία 106 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 107 στη σελίδα 20. 107 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 108 στην επόμενη σελίδα. Συμβαστική τροπολογία 108 με ονομαστική κλίση. την ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 109. Ονομαστική ψηφοφορία. Και εδώ άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45-59. Ή μήπω όχι. Όχι, λάθος. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 110. Συμβαστική τροπολογία 110. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 111 α στη σελίδα 23 με ονομαστική κλίση 110α τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 111 σελίδα 23 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία συμβαστική 111 Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 112, στη σελίδα 27. Με ονομαστική κλίση. Συμβαστική 112, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην συμβαστική τροπολογία 113 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 114 στην επόμενη σελίδα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 115. Στη σελίδα 29. Συμβαστική τροπολογία 115 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 116 στη σελίδα 31. Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 4715 του κυρίου Αρντός. 4715 υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 118 με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 119 με ονομαστική κλίση. «Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4722. Χόιμπουχ. Και Χόισλινγκ. 4722. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 83 Δεύε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84 Δεύε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 120. Μαρμαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 121. Ονομαστική ψηφοφορία και εδώ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 122. Στη σελίδα 35. Άρχεται ψηφοφορία ονομαστικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 48, στην τροπολογία 4800. Σελίδα 36. Τροπολογία Χόισλινγκ Χόιμπουχ. Ποιο είναι υπέρ τη 4.800. Κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 123. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 124, στη σελίδα 37, με ονομαστική κλίση. 124 συμβαστική τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Στη σελίδα 38 ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 125 με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία, τέλος ψυχοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 126, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψυχοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 127, με ονομαστική κλίση, Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε την τροπολογία 4883 της κυρία Ζωανά και τροπολογία 59 της Επιτροπής Γυναικών. Ταυτόσημη. Υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 48, 83 και 59. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Κομπρόμις 120. Τροπολογία συμβαστική 129 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 130 στην επόμενη σελίδα. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 131. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 132, ονομαστικά άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4907. 4907. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 4908 υπέρ εγκρίνεται 4909 υπέρ κατά απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία 135 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 138 ονομαστικά Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4918 του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 140 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 141 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 415 της Συγγήτριας που καλύπτει και την 213 της Ρέτζη. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. Είμαστε εντάξει. Τελειώσαμε με αυτή τη σελίδα, με αυτό το κατάλογο. Πάμε στο επόμενο τμήμα, στα παραρτήματα. Θέλετε, παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή και πάμε στην συμβαστική τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία παραρτήματα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εναλλακτική συμβαστική τροπολογία στη σελίδα 11. Στη σελίδα 11 εναλλακτική συμβαστική τροπολογία με ονομαστική κλίση και αυτή. Εναλλακτική συμβαστική τροπολογία. άρχιτη ψηφοφορία. Ονομαστικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Συμβαστική τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 442. Ναι, στη σελίδα 21, τροπολογία 442. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Ναι. Τροπολογία 442, πρώτη τελευταία σελίδα του συγκεκριμένου, κατάλογου, του συγκεκριμένου εγγράφου. Τις συγκεκριμένες ποιος είναι υπέρ της 442, εγκρίνεται. 443 και πάλι τις συγκεκριμένες ποιος είναι υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 443 της ηγήτρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 444 της ηγήτρια. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 52-45 Νέκοφ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ή δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε στην 445 της ηγήτριας. 445. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 446 υπέρ. Εγκρίνεται. 447 της ηγήτριας και πάλι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 240 της Ρέτζη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 448 της Σιγήτριας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 199α της Έμβη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 199 β της έμβη. Όχι, πρώτα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 199 α της έμβη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται. 199 β έμβη. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 200 της έμβη, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 200 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5248 του κυρίου Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και πάμε στο τελευταίο έγγραφο. Το κατάλογο ψηφοφορίας για τις αιτιολογικές σκέψεις. Και πάμε τροπολογία 1 στη σελίδα 2 της Επιτροπής Ρέτζη. Ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 1 στη σελίδα 2, Επιτροπή Ρέτζη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 471. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 469. Ή μάλλον 477. Τι γίνεται. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Τώρα με ενημέρωσαν. 5.49. Στη σελίδα 8, στη σελίδα 8, 5.49, Χόιμπουχ και Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 7 της υπέρ. Εγκρίνεται. 8 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 8 της ΔΕΒΕ τέλος ψηφοφορίας 8 της ΔΕΒΕ τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται πάμε σελίδα 9 τώρα 569 τροπολογία του κυρίου Ροπέ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 572 και 19 υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στην 571 και 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτονται. 13 της έμβη υπέρ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 591. Α, συγγνώμη, ζήτησα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 570 παρακαλώ, αλλά βιαστήκατε λίγο. Θα ήθελα ηλεκτρονικό έλεγχο για την 570. Ναι, αλλά προηγουμένω είχαμε την 569. Και από τη στιγμή που εγκρίθηκε έπρεπε να πάμε κατευθείαν στην 571. Δεν χρειάστηκε καν να ψηφίσουμε. Την 570 κατέπεσε. Εντάξει. Πάμε στην 591, Χόισλιν και άλλων. Και υπό παράγραφος 1. Ποιος είναι υπέρ και 11 της Ρέτζη. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία για την 591. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 της έτσι. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 έμβη. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 592 του κυρίου Νέκοφ. Υπέρ. Εγκρίνεται. 13 πρώτο τμήμα της ΔΕΒΕ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 593. Μαγκίνες, υπέρ. Εγκρίνεται. 594. Υπέρ. Εγκρίνεται. 595. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 595. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 5.96. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5.91. Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 608 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 599 και 600 υπέρ. Εγκρίνονται. 598 υπέρ. Ή μάλλον 597 597 του κυρίου Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Με αυτό είπα και εγώ. Πάμε στο 597 του κυρίου Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 603. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 604. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 604. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 606. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 601 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 δεύτερο τμήμα. Ντέβε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 Ρέτζι. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την τροπολογία 11 της Επιτροπής Ρέτζι. Δεύτερο τμήμα. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 της ΕΜΒΗ. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογίες 609 και 6. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 612 και 613. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 16. Ή μάλλον πάμε κατευθείαν στην 14 της ΔΕΒΕ 15 λέει ο πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ. 15, 15. Κατά. Απορρίπτεται. 622 και 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 623 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 623. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 624. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 624. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 625. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της ΔΕΒΕ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 16 της ΔΕΒΕ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Δεν σηκώνω τα χέρια σε 626. 626 Χόισλινγκ και άλλων. Ποιο είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 της ΕΜΒ, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Με μία ψηφοδιαφορά απορρίφθηκε. Τροπολογία 20 της ΕΜΒ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 627 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως για την 627. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 της ΔΕΒΕ. Άρχεται ψηφοφορία. Ε, ποιος είναι υπέρ, συγγνώμη, κατά. Απορρίπτεται. 633 της κυρίας Νόιχλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία, στη σελίδα 19. Τροπολογία 705 του κυρίου Κάρθη. 705. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Στη σελίδα 22 τώρα, τροπολογία 738, 738 και 29. Ποιος είναι υπέρ του κ. Γιακόφτσιτς. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Πάμε στην τροπολογία 776 του κ. Νταντά. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 779 του κυρίου Χόισλινγκ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Μαζί με την 25 της Ντεβε. 782 Σένρα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 785 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28 και 788. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Πάμε στροπολογίες παρακάτω, φιλομετράμε υπομονετικά, στη σελίδα 32, τροπολογία 893 και 894. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 23 της Ρέτζη, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 892, 895. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 895. Νόιχλ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 907. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 910 και 911. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 910 και 911 έρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 909. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 908 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 913 υπέρ κατά απορρίπτεται 914 υπέρ κατά απορρίπτεται κρίμα 915 και 916 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 919 υπέρ. Ή μάλλον λάθος, λάθος διορθώνει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, 917, 917. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 919. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 919 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 920. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 918 υπέρ κατά απορρίπτεται 912 υπέρ εγκρίνεται 39 της έμβη υπέρ κατά απορρίπτεται 26 ρέτζι υπέρ κατά απορρίπτεται 927 και 928 υπέρ κατά απορρίπτονται Τροπολογία ηλεκτρονικός έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία 927 και 928. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτονται. 27 της Ρέτζι Περ. Εγκρίνεται. 942. Δελαέ και Νταντάν. Ποιος είναι υπέρ. Σελίδα 34. Εγκρίνεται. 951. 951. Νόιχλ και άλλων. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Καλύτερα για την 951. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 969 ε, για τον κανονιστικό υπερθεματισμό. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ των προπολογισμών. Εγκρίνεται. 974. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 975. Υπέρ. Είμαι 975. Υπέρ. Εγκρίνεται. 972 και ή μάλλον όχι, όχι. Μια και εγκρίθηκε η, προ... η 975, πάμε στην 971, 970 ε, και 971. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. 978 του κυρίου Μέλου, υπέρ. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 31. ΔΕΒΕ 31 που είναι Πάμε στην 998 του κυρίου Νέκοφ. 998 Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Σελίδα 40 στο δικό μου έγγραφο και τροπολογία Τι γίνεται Τι έγινε με τη δερμηνή. Υπάρχει πρόβλημα γερμανικά Εντάξει τώρα. Μάλλον έγινε αλλαγή στους διερμηνείς και χάθηκε για λίγο. Τροπολογία 10.32 Χόισλιν και 34 Δεβε ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 1035 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38 της Ήγητριας υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1033 και 49 υπέρ κατά απορρίπτονται. Τροπολογία 1034 ή μάλλον προηγουμένως θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα για τις τροπολογίες 1033 και τη 49 της ΕΜΒΙ. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 1034 και 32 ρέτζι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 1039 και 15 φαμ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογίες 1037 και 1038. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 12 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1055 του κυρίου Κάρθη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 των προπολογισμών. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1056 του κυρίου Έρντο. Υπέρ. Εγκρίνεται. 1065 του κυρίου Έρντο και πάλι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1068 πάμε. Όχι, όχι, όχι. Συνεχίζουμε κανονικά. 1064. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 και 1066. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 1068. 1068 του κυρίου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 52 έμβη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1070 του κυρίου Κάρθη υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 1071 Τον Λουαζό και Κολομπιέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1073 Εράνς και άλλων υπέρ. Εγκρίνεται. 43 ε, συγγνώμη, 1074 της κυρίας Πετήρ. Ποιος είναι υπέρ. 1074 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη 1074 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η 1074. μπορούμε χωρίς διάλειμμα να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης, όπως έχει τροποποιηθεί. Όχι, ζητάτε διάλειμμα. Καλώς, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα τότε. Κάποιος πρότεινε μια σύντομη διακοπή. Ένα σύντομο διάλειμμα θα κάνουμε, μια και το ζήτησαν οι συνάδελφοι. E, Δεν θέλετε να ψηφίσουμε γιατί πρότεινα κάποιο διάλειμμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τελική ψηφοφορία. Αλλά μια και έχουμε μία μόνο ακόμη ψηφοφορία, δεν χρειάζεται να την αναβάλουμε. Είναι τόσο σημαντική αυτή η ψηφοφορία για τους αγρότες μας, για τους γιώργους και μας που περιμένουν πώς και πώς. Και είναι σημαντικό να δείξουμε έργο, να δείξουμε αποτέλεσμα. Τι αποφασίστε, τελικά, διάλειμμα ή όχι. Όχι. Ψηφίζουμε κατευθείαν. Ο κύριος Νίκολσον. Εγώ προτείνω να γίνει ψηφοφορία τώρα. Καλώς, ψηφίζουμε. Και άλλοι συνάδελφοι προτιμούν να ψηφίσουμε αμέσως. Ο κύριος Δεκάστρο. Συνάδελφοι, καλά ερμηνεύσατε τη σημασία αντίθετης, αντίθεση. Ε, απόρριψη σημαίνει αντίθετη ψήφος. Λοιπόν, προσοχή. Εγώ προτείνω να κάνουμε δύο λεπτά παύση για να αξιολογήσουμε σωστά την ψηφοφορία που θα κάνουμε. Μια δική μας αντίθετη αρνητική ψήφο σημαίνει απόρριψη. E, λοιπόν, ε, ανταλλάξαμε απόψεις. Συνεννοηθήκαμε, ο κύριος Ταραμπέλα λέει να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης για τα στρατηγικά σχέδια όπως έχει τροποποιηθεί. Όπως είπα είναι πολύ σπουδαία αυτή η ψηφοφορία ε, γιατί δείχνει το έργο μας στους Ευρωπαίους αγρότες. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Η κυρία Ράς Γκαρσία, αν κατάλαβα καλά αν απορριφθεί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έκθεση, απορρίπτεται και η χθεσινή και επιστρέφει το σύνολο της δέσμης προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι. Η δική μου απόρριψη θα συμπαρασύρει και τη χθεσινή. Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμότατα. Καταρχήν θερμά ευχαριστώ στην εισηγήτρια που έχει και το λόγο, κυρία Ρας Γκανσία. Ξέρω ότι επίπονο, πόσο επίπονο ήταν το έργο σας, πόσο εργό τις προσπάθειές σας, πόσες χιλιάδες τροπολογίες χρειάστηκε να εξετάσετε και να συνδυάσετε. Κύριε Ιακώφτης, καθίστε παρακαλώ κάτω, δεν βγαίνουμε ακόμη από την αίθουσα. Ας ακούσουμε την εισηγήτριά μας, την κυρία Ράς Γκαρσία. Μη σηκώνεστε παρακαλώ, καθίστε. Κυρία εισηγήτρια έχει το λόγο. η συγκίνηση, η συγκίνηση είναι η αιτία. Από τη συγκίνηση έχισα το νερό κάτω, έβρεξα τα έγγραφά μου, τα μουσκεψα όλα. Πάντως θα ήθελα να συγχαρώ α, α, θερμότατα τον Ευρωπαϊκό κλάδο τη Γεωργία και τη Κτηνοτροφία. Χάρη στην πρόταση αυτή, τροποποιείται ουσιοδό η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτιώνονται οι προποθέσει και επιτυχάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δίνουμε ενάψματα, κίνητρα στου παραγωγού μα να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο προηγμένες τεχνολογίες, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας για να βρεθούν στην πρωτοπορία όπως ήταν μέχρι τώρα, στα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καλής μεταχείρισης των ζώων και ασφάλειας των τροφίμων. Ευχαριστώ θερμότατα τους συναδέλφους για τη συμπαράστασή τους, την προσπάθειά τους, τη συνεργασία τους. Και τέλος θα ήθελα, θα ήθελα το επόμενο κοινοβούλιο όταν θα ξαναρχίσουμε, θα συνεχίσουμε το έργο μας στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, να ετοιμάσουμε το συντομότερο δυνατό το έγγραφο αυτό για να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αυτό που μας ζητάνε οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μας είναι ασφάλεια δικαίου το συντομότερο δυνατό και ένα κατάλληλο προϋπολογισμό φυσικά. Και Μιλούμε και για τον κατάλληλο προπολογισμό στο έγγραφο αυτό, γιατί αυτή είναι η θέση μα, τη διαφύλαξη των κονδυλίων του γεωργικού προπολογισμού, τη κοινή γεωργική πολιτική. Θερμά ευχαριστώ και βάζω τελεία εδώ. Μάλιστα. Πριν αρχίσουμε τις ευχαριστίες, έχω μία παρατήρηση. Γι' αυτό σας έδωσα την... Ε, ε κρίμα που χύσατε νερό. Θα μπορούσατε σαμπάνια να χύσετε. Ευχαριστώ θερμότατα και εγώ την εισηγήτρια και όχι μόνο τους και ηγητές επίσης, τους βοηθούς και συνεργάτες της ηγήτριας, των σχεδόν εισηγητών, της γραμματείας, όλους τους συντάκτες γνωμοδότησης, όλους όσοι συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτού του εγγράφου. Ξέρουμε πόσες συζητήσεις έγιναν ατέλειωτες συναντήσεις Φυσικά στι συμβαστικέ προτάσει και ο συμβασμό δεν μπορεί να ικανοποιεί του πάντε, αλλά αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του καλή συμβασμού. Αν ήταν συμβασμό που ικανοποιούσε μερικού κάποιο μόνο, δεν θα ήταν συμβασμό αλλά μονόπλευρη ικανοποίηση μια παράταξη. Χαίρομαι λοιπόν που καταφέραμε να συμφωνήσουμε και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπέβαλε την πρόταση, την αρμόδια Γενική Διεύθυνση με τους υπαλλήλους της και να κηρύξω το πέρας της συνεδρίασής μας. Νομίζω ότι ε, αξίζουμε ένα καφεδάκι. Ε, μέχρι το τέλος της θητείας ε, δεν θα προλάβαινα να έπινα αυτό τον καφέ επιτέλους. Αλλά ευτυχώς τελειώσαμε και νωρίτερα μάλιστα, 11.30. Σας ευχαριστώ θερμότατα όλους και τους διερμηνείς. Ποιον, ποιον ξέχασα, ξέχασα κανένα από τις ευχαριστίες. Αρκούν, αρκούν αυτές τις ευχαριστίες. Αν ξέχασα κάποιον, ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να συνεδριάσουμε το απόγευμα. Τώρα η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 8 Απριλίου. Σας κάνω και δωράκι το ελεύθερο απόγευμα, μια και δεν χρειάζεται να συνεδριάσουμε σήμερα το απόγευμα. Ε, περίμενα το χειροκρότημα, μια και σας έκανα δώρο ένα ολόκληρο απόγευμα. Ακυρώνεται η απογευματινή συνεδρία στο επόμενο ραντεβού είναι στι 8 Απριλίου. Γεια σας.